θα διανεμηθούν προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση και αν δεν διαφωνείτε θα διαβιβάσω στους αρμοδίους δικαιούχους και αποδέκτες τα όσα μόλις ψηφίσαμε. Η περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται. Εύχομαι σε όλους τους αδέλφους ασφαλή επιστροφή και αναζωογονητικές θερινές διακοπές. Με